θα αναδειχθεί αυτή η στεναρή θέση του Κοινοβουλίου. Ε, το ελπίζω ειλικρινά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Επίτροπο. Πρέπει να σας πω ότι έχω ε, λάβει δύο ψηφίσματα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση η οποία κλείνει εδώ. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12.30. Η επόμενη συνεδρίαση θα ε, αρχίσει αύριο, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί. Η σε διάταξη έχει ήδη αναρτηθεί